Der Präsident! Vielen Dank. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich Καθίστε κυρίε και κύριοι και κηρύσω την επανάληψη της συνόδου που Διακόπηση 27 Μαΐου, αγαπητοί συνάδελφοι. πρώτο ξεκινήσουμε τις εργασίες μας.